να εγκριθεί ε, κατά την επόμενη θητεία. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό δεν μπορεί να γίνει ήδη τώρα, αλλά ελπίζω να αρχίσουμε τους τριμερείς διαλόγους κατά τα ε, τέλη Σεπτεμβρίου. Όλοι είμαστε δεσμευμένοι να έχουμε μια Ευρώπη που προστατεύει και που κάνει τους πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο και εγώ ε, σας ε, καλώ να στηρίξετε αύριο τα σημαντικά στοιχεία αυτής της νομοθετικής πράξης και με τον τρόπο αυτό θα κλείσουν τα κενά ασφαλείας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς το να έχουμε μια πιο ασφαλή Ευρώπη για όλους μας τους πολίτες. Και τώρα επιτρέψτε μου να απαντήσω στον συνάδελφο συνάδελφό τον κύριο Μαριά, στα ελληνικά. Σημαντικό θέμα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ερώτησή σας δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα. Επειδή όμως συμμερίζομαι την ευαισθησία σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου στείλετε μια έγγραφη ερώτηση. Θα φροντίσω να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες, να πληροφορηθώ και να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο εισηγητής κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ αυτό και θέλω να πω ότι για μένα και για το ΕΛΚ το να παραμείνει το σύστημα είναι καθοριστική σημασία. Αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, το σύστημα θα χάσει, ε, δεν θα προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ε, αν αφαιρέσουμε αυτό το σύστημα. Ως εκπρόσωπος των ε, πολιτών, εκπρόσωποι όλοι μας πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους. Είμαστε υπόλογοι έναντι των πολιτών για το ότι διεκδικούμε την ψήφο τους και είναι σαν σαφές ότι όλες οι απόψεις είναι νομιμοποιημένες, αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτοί που πιστεύουν ότι το θέμα αυτών των θεωρήσεων ε, που πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και εκείνοι που πιστεύουν ότι ε, πρέπει να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά, όλοι αυτοί πρέπει να εξηγήσουν τις απόψεις τους στους ψηφοφόρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και συγκητέ για την προσφορά τους, να ευχαριστήσω επίση τους συνεργάτες, τις γραμματείες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί όλοι σας ήσασταν καθοριστικοί για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Ντάλη με θέμα θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Το λόγο έχει η συγγήτρια, κυρία Ντάλη, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις για τη συνεισφορά τους. Είχαμε πληθώρα συζητήσεων για τις ευρωπαϊκές αξίες, την αρχή της αλληλεγγύης καθώς και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους και να λάβουμε αποφάσεις ακόμα και αν δεν είναι δημοφιλείς. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ασχοληθήκαμε με το μεταναστευτικό. Θεωρήσαμε ότι θα λυθεί από μόνο του. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι' αυτό πολλοί απογοητεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάθηκαν και ζωές. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να εργαστεί πολύ σκληρά για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε προς ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Το ζήτημα όμως μπλοκαρίστηκε σε επίπεδο Συμβουλίου εδώ έχουμε ένα ταμείο 10 δις, το οποίο συστάθηκε και τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Το θέμα της ε, μετανάστευσης δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εκτός συνόρων μας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται αρρωγή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ε, δυσκολίες που υπάρχουν και είναι αντικειμενικές. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ προέρχομαι από τη Μάλτα, μια χώρα που γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Σώσαμε ζωές, δεχτήκαμε πολύ κόσμο και δείξαμε αλληλεγγύη. Υπάρχουν και άλλες χώρες που αντιμετώπισαν το ίδιο ζήτημα και το γνωρίζει πολύ καλά ο Επίτροπος. Μιλάμε για μία αρχή, την αρχή αλληλεγγύης που διέπει το έργο αυτού του ταμείου. Στις πόλεις υπάρχει συνεργασία με τις περιφέρειες, κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ για να ελαχιστοποιήσουμε τον φόρτο της παράνομης μετανάστευσης. Επίσης έχουμε και ασυνόδευτους ανηλίκους θα πρέπει να τύχουν ειδική μεταχείρισης. Ο τίτλος του Ταμείου αφορά την συγχώνευση, την ένταξη αυτών των ανθρώπων στον ε, κοινωνικό ιστό. Υπάρχουν ε, τέσσερα δις για τη συνδρομή ευρωπαϊκών κρατών που βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή του ζητήματος. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη δυνατή χρήση αυτού του ταμείου γιατί είναι το μόνο εσωτερικό ε, μέσο, η μόνη εργαλειοθήκη που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στα εσωτερικά μας σύνορα. Θα πρέπει να έχουμε στοχοθετημένη εργασία και το Ταμείο αυτό θα πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τρίτες χώρες. Δεν θεωρούμε ότι θα μπορέσει να υποκαταστήσει βεβαίως άλλα ταμεία. Μας απασχολεί και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης καθώς και της ένταξης και αλληλεγγύης. Αυτές οι ελάχιστες ποσοστίες αναλογίες εντάσσονται εδώ για να υπάρχει ευελιξία, αλλά κάθε στόχος είναι αυτοδύναμος για να μην μείνει πίσω καμία χώρα. Κάθε χώρα θα πρέπει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Εάν ισχύει η αλληλεγγύη που λέμε, αναφέρουμε εδώ και πέντε χρόνια, εάν πραγματικά ισχύει, θα πρέπει τότε η, ο λόγος να γίνει δράση. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Θα ήθελα να πω ότι απόψε Θα ήθελα να αρκεστούμε στον χρόνο, ε, στον χρόνο μιλίας, γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε στα μεσάνυχτα. Γι' αυτό να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ντάλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τον γρήγορη εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προπαρασκευή των τριών εκθέσεων για του τρει σημαντικού αυτού φακέλου που θα συζητήσουμε απόψε, και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευση. Πολλά από τα σημεία που θα αναφέρω είναι οριζόντια φύσεω και αφορούν και τα τρία ταμεία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ελπίζω το Συμβούλιο σύντομα να εγκρίνει και την διαπραγματευτική εντολή. Η μετανάστευση και η ασφάλεια εξακολουθούν να είναι από τις πιο σημαντικές ανησυχίες των συμπολιτών μας σήμερα. Χρειαζόμαστε επαρκείς πόρους για να υποστηρίξουμε τις δράσεις μας στον τομέα αυτών, σύμφωνα με τις πολιτικές μας προτεραιότητες και συμπληρωματικά με, τα, με όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτή τη στιγμή δίδεται ενίσχυση σε ένα εκατομμύριο τούντες άσυλο αυτή τη στιγμή. και 3,5 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτου χωρών λαμβάνουν υποστήριξη για ένταξη. Τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, να, δεν να έχει επιτευχθεί χωρί την βοήθεια του κοινοτικού προπολογισμού. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να εξελιχθούν και η χρηματοδότησή μα πρέπει να είναι ευέλικτη, να είναι απλοποιημένη και να μπορεί να προσαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ενίσχυση του συνολικού προπολογισμού για τη μετανάστευση τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια πάνω από 36 δις για την περίοδο 2021-2027 από τα οποία 10,4 δις για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Αυτό καταδεικνύει την πολιτική σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καλύτερη διάγηση της μετανάστευσης, των συνόρων και των προκλήσεων για την ασφάλεια. Γνωρίζω ότι συμμερίζεται αυτή την άποψη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης πιο συγκεκριμένα θα υποστηρίξει την ενίσχυση της, του κοινού συστήματος ασύλου της Ευρώπης, την νόμιμη μετανάστευση στα στα μελη και υποστήριξη για την ένταξη σε ό,τι φορά του τρίτων χωρών. Στα πλαίσια των στόχων αυτών θα δοθούν και κίνητρα για μέτρα ένταξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως μαθήματα γλωσσών και μαθήματα ε, αγωγής του πολίτη σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη. Τα ταμεία αυτά θα μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε και την παράτυπη μετανάστευση για την επιστροφή, με την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να παραμένουν στην Ένωση. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε όμως, πέρα από τον αυξημένο προπολογισμό, πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ευελιξία για τα ταμεία μας. Χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά μέσα που θα υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες καθώς αναπτύσσονται έως το 2027. Τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη μας όταν το χρειάζονται. Δεν μπορώ να υπογραμμίσω το θέμα της ευελιξίας. Η ευελιξία σχετίζεται και με τους τρεις αυτούς, τρία, τετρία αυτά τα μία που θα συζητήσουμε, μέσω της θεματικής αυτής διευκόλυνσης και την ενδιάμεση αξιολόγηση μας επιτρέψουν να διαθέσουμε 60% της χρηματοδότησης με βάση τις εξελίξεις των αναγκών και των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων ε, ανα πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα έχουμε 50% χρηματοδότηση με τα κράτη-μέλη για να υποστηρίξουμε δράσεις και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επίσης έχουμε προτείνει να απλοποιήσουμε απλοποιήσουμε την εφαρμογή, την υλοποίηση. Η διαχείριση των ε, ταμείων θα διευκολυνθεί και θα γίνει πιο απλή μέσω ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων σε ό,τι αφορά τα ταμεία μοιρασμένης διαχείριση. Δημιουργούμε και συνέργεια και συμπληρωματική προσέγγιση σε σχέση με τους στόχους μετανάστευσης και ασύλου στα πλαίσια των διαφόρων ταμείων. Σε τομείς όπως η ένταξη υπηκών τρίτων χωρών, τα μέτρα κατά τη ριζοσπαστικοποίηση, η συνεργασία με τι εταιρού, με τις, χώρες Εδώ η Κομισιόν επιφυλάσσεται για την ώρα βέβαια, αλλά πρέπει να πούμε ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θέτει κάποια εμπόδια σε ό,τι αφορά την ευέλικτη χρήση των ταμείων και εμεί δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Τα ελάχιστα ποσοστά δαπανών αποτελούν εμπόδιο για την ευελιξία. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ανάγκες και εμπειρίες, ε, έχουν άλλα επίπεδα πίεσης. Θα πρέπει να μπορούμε να στείλουμε τη χρηματοδότηση εκεί όπου χρειάζεται. Επιπλέον, η πρόταση αυτή θα καταστήσει αυτά τα ταμεία ακόμα λιγότερο ευέλικτα από στο παρελθόν και θα προσθέσει βεβαίως ε, διοικητικό άχθος και άχθος εποπτείας η δημιουργία ισχυρών ε, συμπράξεων με τις χώρες προέλευσης και τράνζιτ είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη στιγμή. Η στενή συνεργασία με τους εταίρους μας είναι ένα ζήτημα κλειδί για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι ε, προκλήσεις αυτές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όλος ιδιαίτερω τα εξή. Η δημιουργία ενός μέγιστου ορίου για τις εξωτερικές δράσεις και να, και να δεχόμαστε τη συνεργασία μόνο σε ειδικέ περιπτώσει δεν θα επηρεάσει μόνο την ευελιξία του Ταμείου, αλλά και την επίτευξη των στόχων ασφάλεια και μετανάστευση τη Ένωση. Επιπλέον, έχουμε προτείνει ε, πολύ αυστηρέ προποθέσει, 30% απορρόφησης από τα κράτη-μέλη για να μπορούν να έχουν περαιτέρω χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμα. Και υπάρχουν και στοιχεία αυστηρότητας και συστηματική διευκόλυνση μέσω πράξης και κατεξιοδότηση, κά, κάτι που δεν γίνεται και νομικά. Είναι πιο σημαντικό λοιπόν από ποτέ ε, να έχουμε μια σωστή, σωστό σχεδιασμό ε, των εργαλείων μας που θα μπορούν να αντέξουν στο χρόνο. Ε, ευχαριστώ κυρία Αβραμόπουλε και τώρα θα δώσω το λόγο στην Έλλη Σλάιν που θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστώ κυρίω την εισηγήτρια, την κυρία Ντάλη, για τη δουλειά που έκανε σε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω και του συναδέλφου τη Επιτροπή Ανάπτυξη, με του οποίου προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια νέα εξωτερική διάσταση του Ταμείου που θα λαμβάνει υπόψη τη ε, τι επιπτώσει σε τρίτε χώρε και να μην επιβληθούν, ε, χωρί να είναι σωστό, ε, συγκεκριμένε απόψει που θα οδηγήσουν υποτίθεται στο να εξαλείψουν την φτώχεια. Η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι μια πολύ καλή είδηση. Να υπάρχουν βέβαια τα απαραίτητα κονδύλια για να προάγουμε την ενσωμάτωση, την νόμιμη διαβίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εργαλείο αυτό δεν πρέπει να τύχει εκμετάλλευση για να γίνουν περαιτέρω επαναπροωθήσεις γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις επιπτώσει στην χώρα από την οποία προήλθαν οι ε, μετανάστες. Το θέμα της Λιβύης, πράγματι αυτό πολύ σωστά θίγεται και αυτό που έχει σημασία είναι, όπως σας είπα, να υπάρχει νόμιο δόσης ε, για τους ε, μετανάστες. Ευχαριστούμε την κυρία Σλάιν, επόμενη μιλήτρια από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ο κύριος Ντανιέλε Βιώτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πάνω από 10 δισεκατομμύρια κατά τα επόμενα έτη. Ε, αυτό θα πρέπει είναι το σημείο κίνηση για να υπάρχει σαφώ μια κοινή πολιτική ασύλου και ενσωμάτωση που θα βασίζεται στι αρχέ τη αλληλεγγύη. Οι μεταναστευτικέ ροέ, όπω ξέρουμε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που απαιτεί και μια νέα απάντηση από την Ευρώπη. Ε, θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ιταλία, το οποίο όμως το ακυρώνει ο κύριος Σαλβίνη με ένα διάταγμα που θα φέρει μόνο ανασφάλεια. Ε, κατά την άποψη της Ιταλίας και του κύριου Σαλβίνη ε, θα πρέπει να βρεθούν ε, υποτίθεται μακροπρόθεσμες λύσεις για την μετανάστευση αλλά κύριε Επίτροπε δυστυχώς έχουμε πλέον τις λαϊκιστικές δυνάμεις που έχουν την κυβέρνηση στην Ιταλία και αυτοί επιθυμούν να αφήσουν ανοιχτό το θέμα των μεταναστών για να κάνουν μια αέναη και συνεχή προεκλογική εκστρατεία. Στο και θα έλεγα. Για δέστε λοιπόν σήμερα την αίθουσα. Ούτε ένας εκπρόσωπος από την Ιταλία, ούτε ένας εκπρόσωπος από την πλειοψηφία στη χώρα μας που θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί εδώ για να συζητήσουν τα προβλήματα. Εγώ κύριε Επίτροπε σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστώ και εσάς και την κυρία Ντάλη. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο Βιώτη και τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, εκ μέρους του ΕΛΚ, ε, ο κύριος Λένερς. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η μεταναστευτική κρίση είναι μία από τις βαθύτερες κρίσεις στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα τελευταία χρόνια ένα πράγμα κατέστη απόλυτα σαφές, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μας απάντηση. Αυτό το νέο ταμείο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ κύριε Βραμόπουλε που προτείνετε να τριπλασιαστούν τα κονδύλια αυτού του ταμείου. Το έχει ζητήσει αυτό το ΕΛΚ και χαίρομαι πάρα πολύ που η Κομισιόν θα το κάνει. Όμως για να σημειώσουμε ουσιαστικά αποτελέσματα αποτελέσματα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο ε, επαρκή πόρους, χρειαζόμαστε και ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Να υπάρχει και ισορροπία όσον αφορά τους στόχους του Ταμείου. Κατανοώ βέβαια κάπως ε, την απογοήτευση που νιώθει ο κύριος Επίτροπος, ε, την διέβλεψα στην ομιλία του, γιατί από ό,τι φαίνεται η αρχική πρόταση κάπως μέχρι το τέλος έχει χαθεί, έχουν χαθεί πολλά τη στοιχεία. Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας βασίζεται στη νόμιμη νόμιμη, νομότυπη μετανάστευση, ενώ δεν γίνεται κανένα λόγο, σχεδόν κανένα λόγο για την αντιμετώπιση τη παράτοπης μετανάστευση. Θα έπρεπε, παραδείγματο χάρη, ε, να επισημάνουμε ότι προβλέπονται κονδύλια για πάρα πολλά εκτό από την παράτυπη μετανάστευση. Και ο κύριο Επίτροπο το είπε. Αν όμω θέλουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση, πρέπει να συνεργαστούμε και με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, με χώρε προέλευση και διέλευση. Αυτό είναι καθοριστικό στρατηγική σημασία. Δυστυχώ, οι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστούν σχεδόν αδύνατο να συνεργαστούμε με τρίτε χώρε επί των θεμάτων αυτών. Είμαι απογοητευμένο που η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η αντιμετώπιση τη παράτυπη μετανάστευση και η ε, επιστροφή των παράτυπων υπηκών τρίτων χωρών, ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. Όχι, για μα, για το ΕΛΚ, είναι σημαντικό. Όλοι οι μεγάλοι στόχοι του Ταμείου είναι είναι σημαντική και γι' αυτό εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογίες για αύριο για να έχουμε ένα πιο ρεαλιστικό ταμείο και θέλω να απευθυντώ σε όλους τους συναδέλφους που έχουν αυτή τη ρεαλιστική άποψη να μας στηρίξουν αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λένερς. Η επόμενη ομιλήτρια από τους σοσιαλιστές η Σεσίλ Κιέγκε Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, για την εργασία σας. Η επιτυχία διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών βασίζεται στις ε, πολιτικές υποδοχής. Πολιτικές που ήταν αλληλέγγυες με βάση το άρθρο 80 της Συνθήκης. Γι' αυτό αποκαταστάθηκε η φωνή μας, φωνή μίας ολιστικής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Κάτι το οποίο θα προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Απριλίου 2016. Το σύστημα χορήγησης ασύλου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ανηλίκους, τις γυναίκες, τις ευάλωτες κατηγορίες για να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης με καλύτερη ευελιξία, περισσότερη μάλλον ευελιξία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει σωστή χρηματοδότηση που θα αποτελέσει τη θέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κιέγκε. Από το ECR η κυρία Βίμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ. Το ε, θέμα αυτό δεν αφορά μια εμπόλεμη κατάσταση ή την οικονομική ε, δυσχέρεια που υπάρχει, απλώς δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να διαχειριστούμε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Εμείς έχουμε τριπλασιάσει τις ε, πιστώσεις για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Ας δούμε τη σημασία ένταξης αυτών των ανθρώπων. Δεν γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο. Στη Σουηδία έχουμε κάνει μακροχρόνιες επενδύσεις για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό την τελευταία δεκαετία. Κάνουμε πολλές επενδύσεις και λάβαμε υπόψη την ένταξη στον κοινωνικό ιστό και επίσης στα σχολεία εντάξαμε αυτά τα παιδιά. Έχουμε καταργήσει γιορτές για να μην, στα σχολεία για να μην υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος σε παιδιά που έχουν άλλο θρήσκευμα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ολιστικά και βεβαίως να επαναπατριστούν εκείνοι που έχουν ε, έρθει παράνομα. Όσοι έρχονται θα πρέπει να προσαρμοστούν στα δικά μας ήθη και έθιμα. Σκά Κέλλερ από τους Πρασίνους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και γιατί υποστηρίξατε και τη χρηματοδότηση των τοπικών κοινοτήτων, γιατί εκεί οι Ευρωπαίοι πολίτες συνδράμουν. Αυτή είναι η Ευρώπη που χρειαζόμαστε και τα χρήματα εκεί θα πρέπει να μπουν. Όμως είναι αυταπάτη να νομίσουμε ότι άλλες χώρες θα ε, μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα μας, δηλαδή να έχουμε κλειστά κέντρα, για παράδειγμα στην Αίγυπτο. Αυτό ε, οδηγεί σε απομάκρυνση από τις αξίες μας. Δεν ήταν αυτές οι αρχές σύστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη και ας χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για αυτούς που πραγματικά ε, τα χρειάζονται για να μπορέσουμε να συνδράμουμε άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κέλλερ. Από η Μαρτίνα Αντερσόν. Ο αριθμό των ζώων που χάνονται στο Μεσόγειο είναι πραγματικά τραγικό. Η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική, μεταναστευτική Πολιτική τη Ένωση έχει ουσιαστικά επιτρέψει τον θάνατο ε, χιλιάδων μεταναστών στη θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση νύπτει τα χέρια, τα χέρια της ε, για αυτή την, την ανθρωπιστική κρίση. Η Λιβική ακτή εξακολουθεί να, να δέχεται μετανάστες ε, πίσω σε κέντρα όπου ε, εξακολουθούν να σαπίζουν, να τους χτυπούν, να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, κάποιοι μάλιστα δολοφονούνται. Το κλίμακα αυτής της κρίσης ε, έχει να κάνει με την πολιτική ασύλου της Ένωσης που έχει διευκολύνει και την, ε, τα βασανιστήρια πραγματικά ντροπή στο ΕΛΚ και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στέλνουν πίσω του ανθρώπους σε μια ασφαλή χώρα. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση που θα βασίζεται στις αρχές της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος. Κανένα ανθρώπινο ε, Ευχαριστώ την κυρία Άντερσον και τώρα για την EFDD ο κύριος Έθεριτζ, έχετε τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τετάρτη 6 Μαρτίου, ο φραντ Τίμερμανς, ο αξιότιμος συνάδελφός σας, είπε ότι η Ευρώπη δεν ζει πια τη μεταναστευτική κρίση που ζήσαμε το 2015 και το υποστηρίζει αυτό από στατιστικά στοιχεία των ΗΕ Εθνών που δείχνει ότι υπάρχει 81% μείωση στη διέλευση στη Μεσόγειο από το 2015 έως το 2019. Καλό νέο, έτσι. Και ξαφνικά είμαστε εδώ με ένα πακέτο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευση, Άσυλο και μετανάστευση που ο μεγάλο κύριο Τίμωνα είπε ότι δεν είναι και τίποτα σπουδαίο πια. Και πού θα διαθέσουμε τα χρήματα αυτά λοιπόν. Περιλαμβάνει ε, το να δωροδοκούμε τρίτες χώρες για να δημιουργήσουν ε, ε, κέντρα που θα διαθεσουμε τα χρηματα αυτα λοιπον περιλαμβανει το να δωροδοκουμε τριτες χωρες για να δημιουργησουν κεντρα που θα κρατουνται οι μετανάστες να, να στέλνονται ε, μετανάστες υποχρεωτικά σε χώρες της Ένωσης όπου θα μείνουν εκεί ελπίζω ότι τελικά δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τα χρήματα των φορολογουμένων. Και τελικά έχουμε μια οργάνωση εδώ που έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να σταματήσει τη μαζική μετανάστευση και επιπλέον θεωρεί ότι είναι και καλή ιδέα τελικά. Έτσι λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ότι όλοι στο πνεύμα ε, της αλληλεγγύης που ακούμε έτσι συχνά αυτή τη λέξη θα πληρώνεται για να υποδέχεται τους ανθρώπους αυτούς ανεξάρτητα το τι πιστεύουν οι άνθρωποι στις χώρες αυτές, στις χώρες υποδοχής. Βεβαίως όλοι φοβούνται, υποτίθεται, τους απέσιους λαϊκιστές ε, που απλά ακούν αυτό που τους λένε οι εκλογείς. Τέτοια ανησυχία για τη μετανάστευση μετά από αυτά που συνέβησαν και στο Westminster σήμερα πραγματικά πιστεύετε ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν θα, θα, θα, μάλλον θα περάσουν απαρατηρήτα. Έχετε πρόβλημα στο σύνολό της Ένωσης, ε, χώρε στις χώρες της Ένωσης που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1 τρίτο των, ψηφο, των ψηφοφοριών, των, των ψήφων θα πάει σε δυνάμεις εκτός του συστήματος. Εάν έχουμε νέες ε, εκλογές και έχουμε τέτοια ζητήματα, πραγματικά η προοπτική είναι 25, 30, 35% είμαι βέβαιη ότι το, το περιμένετε με ανυπομονησία. Πραγματικά σας προτείνω να πείτε στους συναδέλφους γρήγορα να υπάρξει συμφωνία για το Brexit. Ιδάλλως θα είμαστε εδώ για να σας κυνηγάμε και δεν θα περάσετε καθόλου όμορφα. Ε, ε, Ευχαριστώ τον κύριο Έθριτς και τώρα ο κύριος Λεμπρετό από την ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δημιουργώντας αυτήν τη νέα εκδοχή του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να, να, σε αυτή την τρελή μεταναστευτική πολιτική της. Αυτό το κείμενο είναι πραγματικά καταστροφικό. Θέλει να αφιερώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να οργανώσει την επανατοποθέτηση των μεταναστών και να βρεθούν ε, νόμιμε οδοί μετανάστευση. Θέλει επίση να ενθαρρύνει το διάλογο, το διαπολιτισμικό και το διαθρησκευτικό μεταξύ των κοινωνιών υποδοχή και μετανάστευσης. Ενώ ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τι ευρωπαϊκές μα αξίε, ιδιαίτερα την αξιοπρέπεια των γυναικών απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ. Θέλει επίση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί μαζικά τι ΜΚΟ που οργανώνουν αυτήν την ε, άφηξη των μεταναστών όπως η Open Society του George Soros ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να τις ε, καταπολεμήσουμε ε, χωρίς έλεος. Θέλετε εδώ να προδώσετε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και θα εντοπίσουμε τους ευρωπαϊκούς λαούς για να σταματήσουν. Ευχαριστώ τον κύριο Λεμπρετό. Και τώρα δεν βλέπω τον κύριο Επιτίδιο στην αίθουσα. Οπότε θα δώσω το λόγο αυτής αμέσως στον επόμενο μιλητή. Αγουστίν Διαθντεμέρα από το ΕΛΚ. Έχετε ένα μισό λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ταμείο Μετανάστευση και Ασύλου πρέπει να είναι ένα εργαλείο ευέλικτο για να μπορέσουμε να, να προσαρμοστούμε στι μελλοντικέ ανάγκε των κρατών μελών και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν. Και να, ε, ε βεβαίω να είναι επαρκώς, ε, επαρκές για να μπορεί να αποκριθεί στις ανάγκες αυτές. Θα πρέπει να σεβαστούμε το κεκτημένο ε, τη Ένωση για τη Μετανάστευση, να συντονιστούμε με τι διάφορε προτάσει του πακέτου μετανάστευση και ασύλου και βεβαίω και με τα χρηστικετικά ταμεία για την Αφρική και την ε, ε, Λιβύη πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτέ τι μεταναστευτικέ πιέσει για να πετύχουμε και να, και να σεβαστούμε ταυτόχρονα και τι νομικέ μα υποχρεώσει. Πρέπει όμω και αυτοί να εγγυηθούν ότι τα άτομα που φτάνουν στην Ευρώπη θα ε, λάβουν την κατάλληλη υποδοχή θα μπορούν να έχουν μια διαδικασία έτσι ασύλου δίκαιη και ισότιμη. 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το ταμείο πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση των κοινών εργασιών, τη συνεργασία με τι χώρε προέλευση και τράνζιτ, έτσι ώστε τα άτομα τα οποία αναγκάζονται να φύγουν από τι χώρε του να μην πέσουν σε χέρια εγκληματιών. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου χειροκροτούσαν την καταπολέμηση των διακινητών στους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και τράνζιτ. Όμως, οι προσπάθειες δεν αρκούν για να μπορέσουμε να βάλουμε τέλος αυτή την τραγωδία. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το όργανο πρέπει να εγκριθεί, το εργαλείο να εγκριθεί και να ενισχυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε επόμενο ομιλητή είναι ο Χουάν Φερνάντο Λόπε Ακυλάρ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αβραμόπουλε, βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας ε, μιας ε, λυπηρής πραγματικότητας γιατί μιλάμε για μια κρίση εμπιστοσύνης λόγω του μεταναστευτικού. Δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το δίκαιο σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει τη δουλειά του, υποστήριξε την έκθεση τη συντρόφου μας ε, της ε, κυρίας Νταλή προβάλλοντας ένα ταμείο ασύλου και μετανάστευσης με 10 δις 400 ε, εκατομμύρια. Και αυτό για να δώσουμε μία ε, για να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά το θέμα του ασύλου και του μεταναστευτικού. Δυστυχώς όμως τα κράτη-μέλη δεν ε, τηρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν εφαρμόζουν τις αρχή της αλληλεγγύης. Είναι ευσεβής πόθη όλα αυτά από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Ο Εμίλ Ραντέφ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, αυτό το ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση είναι από τα σημαντικότερα ταμεία στι εσωτερικέ υποθέσει, γιατί εδώ προσφέρεται υποστήριξη ε, στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τι μεταναστευτικέ ροέ. Εγώ χαιρετίζω την αύξηση του προπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια απόδειξη ότι το θέμα της μετανάστευσης παραμένει στην ημερήσια διάταξη και καμία χώρα δεν είναι μόνη της για να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη πίεση. Η Βουλγαρία είναι ε, μια χώρα Πρώτη ε, γραμμής στο θέμα της μετανάστευσης. Δηλαδή, εκεί έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες ε, και ε, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των παράτυπων μεταναστών. 40 περίπου της 100 των πολιτών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν δικαίωμα θα πρέπει να επαναπροωθηθούν. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι η λύση για όλους που θέλουν να έρθουν εδώ για καθαρά οικονομικούς λόγους. Όσοι δεν είναι πρόσφυγες θα πρέπει να επαναπροωθούνται. Ε, το Ταμείο λοιπόν ε, πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράντεφ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σενίντερ Μιούλα για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η βάση της κοινή πολιτικής ασύλου είναι η αλληλεγγύη και η κοινή ανάληψη αυτινών. Και παρότι τους τελευταίους μήνες μειώνει το αριθμός των προσφύγων, ε, το άσυλο και η μετανάστευση παραμένει σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την οικονομική υποστήριξη ε, πέρα από το να προσφέρουμε υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Είναι καθοριστική σημασία να στηρίξουμε τους σημαντικότερους θεσμούς ε, της κοινή πολιτικής ασύλου. Είναι λοιπόν δυστυχές το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει στο να συστήσει μια κοινή πολιτική ασύλου και αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του Συμβουλίου. Παράλληλα, είναι μια θετική εξέλιξη το ότι το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης θα στηρίξει την ενσωμάτωση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς την ενσωμάτωση. Δεν μπορεί κανείς ε, να επιτύχει την ασφάλεια με τείχους και με ε, φράχτες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίτα Μούλα. Τώρα έχουμε έναν ομιλητή για τη διαδικασία διάρκεια, τον κύριο Μαριά. Κύριε Μαριά. Το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση οπωσδήποτε πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σε μια φάση όπου υπάρχουν τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο πρέπει να στηρίξει τις χώρες πρώτης υποδοχής τις χώρες οι οποίες πραγματικά υφίστανται τις μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές εκεί όπου πραγματικά οι κάτοικοι δίνουν μάχη και στηρίζουν την προσπάθεια των χωρών τους να σταθούν όρθιες και ταυτόχρονα να φιλοξενήσουν τους ε, άτυχους πρόσφυγες. όμως βεβαίως έχουμε και πάρα πάρα πολλούς παράνομους μετανάστες οι οποίοι κατακλείζουν αυτή τη στιγμή τα νησιά του αιγαίου και νομίζω ότι ορθώς αναφέρεται στην έκθεση ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στις επιστροφές διότι πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό αποφασιστικά ιδίως για τα νησιά του αιγαίου ιδίως για την ελλάδα όπου έχουμε χιλιάδες παράνομους μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και αυτοί θα πρέπει πραγματικά να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες ήλθαν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαριά. Η Julie Ward έχει ζητήσει και εκείνη τη διαδικασία να μιλήσει στο πλαίσιο διαδικασία ε, Catch the Eye η βελτίωση των οικονομικών ε, πτυχών της ε, πολιτικής για τη μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και γι' αυτό χαιρετίζω την ε, πρόοδο που επιτυγχάνεται με την πρόταση. Η συνάδελφός μου έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στο πόσο σημαντικό είναι να επιτρέπεται στις τοπικές αρχές να διδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση. Αποδίδει σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μια ντροπιαστική στάση έναντι των μεταναστών και των προσφύγων. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξεφύγουμε από αυτή την τάση. Ανησυχώ ιδιαίτερα για την πίεση που ασκείται σε πολλούς εθελοντικά να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Όταν οργανώνονται εθελοντικές επαναπροωθήσεις, οι αρχές πρέπει να ε, διαπιστώνουν ότι πράγματι αυτό είναι δική τους απόφαση. Και αυτό δεν ισχύει σήμερα. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες και οι οργανώσεις της βάσης αναλαμβάνουν ευθύνη για ανθρωπιστική βοήθεια και για την ενσωμάτωση όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ε, έχω μιλήσει πολύ συχνά για την οργάνωση Καλέ και πάρα πολλές άλλες που βοηθούν τους μετανάστες που ζουν στον δρόμο. Ε, λυπάμαι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 12, γι' αυτό θα πρέπει να είμαι αυστηρή ε, και όσον αφορά εσάς κύριε Επίτροπε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά και εσείς πρέπει να ε, τηρείτε τον χρόνο που έχει προβλεφθεί για εσάς. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αβραμόπουλο, ε, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλά μία επιχείρηση λογιστική. Είναι μία σαφή συγκεκριμένη έκφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως προσιλωμένη στο να συνεχίσει να συνεργάζεται με εσά και με το Συμβούλιο για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο στιγμό των δυνατών για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Και ε, ε, προσβλέπω στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, η κυρία Ντάλη, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ και του αδέλφου για τι συνεισφορέ του. Ο κύριο Επίτροπο έχει δίκιο όταν εμένει ότι πρόκειται για μια κρίσιμη βοήθεια για αυτού που τη χρειάζονται. Αυτή είναι και η θέση τη Επιτροπή Ελευθεριών και πρέπει να σα πω ότι το ελάχιστο ποσοστό δαπανών για του βασικού στόχου των πολιτικών μετανάστευση δεν είναι εμπόδιο καθόλου. Στέλνουν τα χρήματα προ του στόχου που έχει θέσει αυτή η Επιτροπή ω προτεραιότητε. Η υποστήριξη της ευελιξίας δεν αποκλείει ελάχιστα επίπεδα χρηματοδότησης για τους στόχους του Ταμείου. Και κάτι άλλο, το να βάζουμε ένα όριο για την εξωτερική χρηματοδότηση εξασφαλίζει ότι αυτό το, το μέσο χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Δηλαδή ένα εσωτερικό χρηματοδοτικό μέσο για την μετανάστευση. Πρέπει να, βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που είναι στην πρώτη ε, γραμμή και κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτό το ταμείο να έρθει να καλύψει κενά από άλλα ταμεία τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και φτάνω τώρα στο, στη δήλωση του ΕΛΚ για τις επιστροφές. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ε, δαπανούν 42% ε, των του κονδυλίου του ε, για τι επιστροφέ, χωρί να υπάρχουν ελάχιστε απαιτήσει. Εξακολουθούν να είναι στόχο των οι επιστροφέ στο Ταμείο. Δεν, έχουν, δεν έχει αφαιρεθεί αυτό και το κράτη-μέλη σίγουρα θα το καταλάβουν αυτό. Δεν είναι βεβαίω ο μόνο στόχο του Ταμείου αυτού. Και βεβαίω ε, η δήλωση αυτή σίγουρα δεν έχει ως στόχο να καταπολεμήσουμε τι καταχρήσει. Προσπαθώ να καταλάβω από πού προέρχεται μια τέτοια ιδέα. Σα ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε ανυπομονησία την ψηφοφορία αύριο. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ντάλη. Και τώρα ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουμε επ' αυτού αύριο. Και τώρα το επόμενο σημείο είναι το πρώτο τελευταίο για απόψε την έκθεση της Τάνια Φαγιών μέσω χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Θα δώσω το λέγω αυτή αμέσω για 4 λεπτά στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω και τα έξι λεπτά μου στην αρχή και θα μιλήσω σλοβενικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις, στις δεσμούς της. Ε, η άνθρωπη των εθνικισμών έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για μια αποτελεσματική πολιτική μετανάστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απελπισία των Ευρωπαίων και των προσφύγων, η έλλειψη αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η αδυναμία να, να φτάσουμε σε κοινέ λύσει είναι κάτι που το εκμεταλλεύονται οι ακροδεξιοί πολιτικοί για πολιτικού λόγου. Αυτό δημιουργεί διαφωνίες, ε, δημιουργεί ε, γαχυποψία μεταξύ πολιτών, μεταξύ κρατών και θέτει σε κίνδυνο το, μέλος της, το μέλλον της, ε, του χώρου Σέγγεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ο, η, η Αυστρία και άλλες χώρες Σέγγεν αυτή τη στιγμή, παρότι έχουν παρ, πάρθει περαιτέρω μέτρα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και παρότι είναι πολύ χαμηλότερος αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη, αυτές οι χώρες για πάνω από τρία χρόνια παρατείνουν ελέγχους στα ιστορικά σύνορα χωρίς αιτιολόγηση. Είναι δύσκολο να εξηγήσω στους ε, συμπολίτε μου από τη Σλοβενία γιατί τους ελέγχουν όταν περνάνε τα σύνορα με την Αυστρία ή τα, τα, τα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας. Θέλουμε ε, ο χώρος της, της Σέγγεν να είναι ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας, χωρί σύνορα. Αυτό είναι που ε, συμβολίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό έχει να κάνει με την σοφία των ηγετών μας, των πολιτικών ηθινόντων. Όμως αυτή η ευθύνη, αυτή η ευαισθητοποίηση φαίνεται να λείπει. Το να έχουμε βεβαίως ασφαλή εξωτερικά σύνορα ε, σημαίνει ότι πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση. Χαίρομαι που συζητούμε σήμερα την πρόταση αυτή, βάσει της οποίας το κοινό ευρωπαϊκό προπολογισμό θα διαθέσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ για τα σύνορα και τις θεωρήσεις. Πρόκειται για το πενταπλάσιο από αυτά που δαπανούνται σήμερα. Είναι πολλά χρήματα εφόσον τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ένα τέτοιο χρηματοδοτικό μέσο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Διότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές έτσι μεταφράζονται σε συγκεκριμένα μέτρα και έτσι μπορούμε να έρθουμε και πιο κοντά στους πολίτες μας. Θα ήθελα όλους ιδιαίτερως να καλωσορίσω το γεγονός ότι υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό 700 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορα μέτρα που αφορούν την Σλοβενία που διαχειρίζεται ένα από τα χερσαία σύνορα της Ένωσης που είναι σε μεγάλη, βρίσκεται σε μεγάλη πίεση ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αυτό το Ταμείο θα βοηθήσει μέτρα σε πρωτοκρατομελών. Έχει δύο πλέον κλειδιά. Το πρώτο είναι μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, έλεγχος των χερσαίων ε, και θαλάσσιων συνόρων, καθώς και κοινέ επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Επίσης, πρόληψη της παράνομης διέλευσης, καταπολέμηση του εσωτερικού εγκλήματος και εφαρμογή του συστήματος πληροφοριών των συνόρων για τον έλεγχο των αγαθών και των επιβατών. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο επιπλέον θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Από το συνολικό κονδύλιο 60% ε, των χρημάτων θα διατεθούν στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών και 40% αφορά μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από την Ένωση. Αυτό το εργαλείο εξασφαλίζει χρηματοδοτική υποστήριξη για, την, για πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη και την δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών, καθώ και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη. Κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι τουλάχιστον 20% των χρημάτων αυτών θα διατεθούν στην πολιτική θεωρήσεων και στην διευκόλυνση τη διέλευση των συνόρων για τους ε, ε καλόπιστους ε, ταξιδιώτες που δεν αποτελούν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η Σέγγεν και είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες αλλά και για τις εταιρείες. Η Σέγγεν είναι επίσης από τα πιο βασικά μέσα έτσι ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να αντιληφθεί τις θεμελιώδεις ε, ελευθερίες του, ελεύθερης κυκλοφορίας ε, και για να μπορέσει να ανθίσει η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά. Επίσης υπάρχουν συστήματα θεμελιών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εφαρμόζοντας έξυπνες τεχνολογίες ενημέρωσης και συνοριακά συστήματα υπάρχει μεγαλύτερο φόβο ε, για την ε, παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Επίση ενισχύουμε τι διατάξεις εκείνες που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά να σέβονται το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιαίτερα την αρχή της απαγόρευσης ε, της ε, ε, Σε ό,τι αφορά τώρα τα hot spot, μπορέσαμε να βελτιώσουμε το σεβασμό της διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προστασίας των ευάλωτων ομάδων μεταξύ των οποίων και τα παιδιά. Αυτό το ταμείο που συζητούμε σήμερα είναι από τα εργαλεία κλειδιά για να υποστηρίξουμε την ε, εφαρμοστική πολιτική της Ένωσης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το ταμείο αυτό, τα χρήματα αυτά που θα διατεθούν τα επόμενα 7 χρόνια, δεν πρέπει να πάνε στη χρηματοδότηση προγραμμάτων σε τρίτες χώρες η διαχείριση των συνόρων της Ευρώπης δεν σχετίζεται με τη δημιουργία ε, κέντρων κράτησης σε τρίτη χώρα ή διατέθοντας το διαχείριση του, του σε τρίτες χώρες. Για να ενισχύσουμε την διαφάνεια τέλος, προτείνουμε ο κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν πιο ενεργά κατά την προπαρασκευή των εθνικών προγραμμάτων. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να παίξει ένα ρόλο παρακολούθησης για να αποφύγουμε οποιασδήποτε υπόνοιες για το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Φαγιόν και τώρα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Φαγιόν, ήδη έχω υπογραμμίσει στην πρώτη συζήτηση που είχαμε ορισμένα οριζόντια ζητήματα που αφορούν και τα τρία ταμεία. Την ανάγκη ευελιξίας και τις συνέργειες με τα άλλα ταμεία και πιστεύω το Συμβούλιο σύντομα θα εγκρίνει την εντολή διαπραγμάτευσης ε, έχει ύψιστη σημασία η χρηματοδότηση αυτή για να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ήδη τέσσερα χρόνια μετά το Π, μπορέσαμε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Έτσι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις μείζονες μεταναστευτικές ροές στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν με βάση τις προκλήσεις και απρόβλεπτα στα σύνορα μας. Επίσης, χρειάζονται συνέργειες με άλλες δράσεις, ευρωπαϊκές δράσεις, για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη ε, δράση μας επιτόπια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ε, τη σύσταση ενός ξεχωριστού ταμείου για τη διαχείριση των σύνορων και την ενίσχυση της ε, σύνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής. Έτσι θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στους ε, τελωνιακούς ελέγχους για να εφαρμοστούν και οι τελωνιακές συμφωνίες και παράλληλα αυτό το μέσο θα χορηγήσει οκτώ δις για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την υποστήριξη της ε, κοινής πολιτικής θεωρήσεων και για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα συστήματα πληροφοριών και να τα επικαιροποιήσουν. Αυτό σημαίνει ε, αύξηση επί τρία των πόρων που προβλέπονταν μέχρι τώρα και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, για να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι τάχιστα σε περίπτωση συνεργειών. Επίσης, η μεγαλύτερη ευελιξία αυτού του μέσου θα βοηθήσει την επιτόπια χρηματοδότηση όπως ε, όσο αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Χρειάζεται μια εύρωστη προσέγγιση ως προς τη διαχείριση συνόρων σε συνεργασία με τις ε, τελωνιακές αρχές. Αυτό το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης θα το κάνει αυτό. Επίσης, ένας άλλος πυλώνας είναι η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει ε, να μπορέσουν οι αρχές των συνόρων να ε, συνεργαστούν με τρίτες ε, χώρες για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και για να μην χάνονται ζωές στη θάλασσα. Θα υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας με τα άλλα μέσα ενίσχυσης των εξωτερικών σύνορων. Έτσι, με τη χρηματοδότηση αυτή θα προωθήσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ε, διαφορετικά, δεν θα μπορέσει να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα που την απασχολούν πολύ περισσότερο. Περιμένω να ακούσω και τη δική σας συμβολή. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κούκαν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία την κυρία Φαγιόν για την πάρα πολύ καλή δουλειά τη. Ω εισηγητή τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εγώ στήριξα αυτόν τον κανονισμό και ζήτησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο σε θέματα διαχείριση. Ζητάμε το ΕΛΚ να τοποθετείται ε, σε θέματα χρηματοδότηση που αφορούν αυτό το εργαλείο, το οποίο έχει ω στόχο να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία αναφέρεται όμως κυρίω στο να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Εδώ λοιπόν χαιρετίζω την αύξηση των πόρων προς το εργαλείο που μεταξύ άλλων θα πρέπει να δώσει σημασία στην ποιότητα της διαχείρισης των πόρων, στις δαπάνες και στην αξιολόγηση. Θέλω να πω ότι είναι επιτακτική ανάγκη το Ταμείο αυτό να συμπληρώνει άλλα εξωτερικά χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαλεία με εξωτερική διάσταση. Επίσης πρέπει το εργαλείο αυτό να συμβαδίζει με θεμελιώδη δικαιώματα και με νομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούκαν και τώρα έχει το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών η κυρία Χολμάια για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια ε, πολύ καλή αλλά και συνεπή έκθεση όσον αφορά το, τη μελλοντική Frontex. Εγώ έτσι θα τη λέω. Έτσι θα τη λέω γιατί είναι και η πιο ε, αποτελεσματική και συνοπτική διατύπωση. Αυτή η αρχή διαχείριση εξωτερικών συνόρων χρειάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε ένα κοινό σχέδιο και ε, είναι επίσης ε, σημαντικό να πούμε ότι πρέπει ως ε, Επιτροπή Προεπολογισμού να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διατεθούν οικονομικοί πόροι για το μέλλον, κυρίως για το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος. Αυτά όλα στο πλαίσιο του πολιτού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που θα υπάρχει νομική βάση έτσι ώστε εκείνα τα οποία μας ενώνουν να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε από κοινού να προωθήσουμε θέματα ασφάλειας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χόλμαερ και τώρα έχει το λόγο ο... οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος ε, Κάρλος Κουαλιού. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Τάνια Φαγιόν για την εξαιρετική μας συνεργασία και να υποστηρίξω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ασφάλεια και την πολιτική θεωρήσεων. Για την επόμενη ε, δεκαετία θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά αυτό το ταμείο. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα οι χώρες που βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή και αυτό αφορά και την ε, σύνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή. Μιλάμε για δέκα δις περίπου. Ε, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Το παρελθόν μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη και άμεση ανταπόκριση. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης. Καλύτερη δικαιοσύνη επίσης.